Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε καλώς ορίζοντας τον εξοχότατο Ιμπραχήμ Αλτζαφάρη, Υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ. Τον συνοδεύει η προσωπία του Γνωρίζετε ότι το θέμα που θα συζητήσουμε είναι το Νταέσ, το Ισλαμικό κράτος και η καταπολέμησή του. Όπως θα ξέρετε, εδώ και μερικές μέρες έχει ξεκινήσει μια μεγάλο διαστάσεων στρατιωτική επιχείρηση. Πού στοχεύει. Στην απελευθέρωση της Μοσούλ. είναι μια πολύ περίπλοκη στρατιωτική επιχείρηση που θα πάρει το χρόνο της. Ας ελπίσουμε ότι το ανθρώπινο και ανθρωπιστικό κόστος που σε κάποιο βαθμό είναι αναπόφευκτο θα είναι όσο μικρότερο γίνεται. είναι δυνάμεις του Ιρακινού στρατού και της εθνικής αστυνομίας που συμμετέχουν και μόνον. Ας ε, είμαστε προετοιμασμένοι με βάση και την πείρα μας από προηγούμενες επιχειρήσεις για να, να αντιμετωπίσουμε τις ε, ανθρωπιστικές συνέπειες αυτής της επιχείρησης. Κύριε Υπουργέ, θα σας δίνουμε το λόγο για την παρουσίαση του θέματος και μετά οι συνάδελφοί μου θα σας υποβάλουν ερωτήσεις. السلام عليكم ورحمة الله جميعا أرحب بكم جميعا أجمل الترحيب في هذا اللقاء Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συνεδρίαση. Είμαι παρόν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το χώρο των λαών, όπου αντυχεί η φωνή των λαών και εδώ θέλουμε να αντυχήσει και η δική μας η φωνή προς όλους τους λαούς του κόσμου. Τα κοινοβούλια είναι το βήμα που επιτρέπει να ακουστεί η φωνή του λαού μας τα κοινοβούλια ψηφίζουν και ελέγχουν τις κυβερνήσεις που κατευθύνουν την εργασία των κυβερνήσεων ανάλογα με τα συμφέροντα των λαών. Το κοινοβούλιο είναι η έκφραση της βούλησης των λαών. Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των λαών. Υπάρχουν βέβαια πολιτικές διαφορές, αλλά οι λαοί είναι όλοι ο ένας στο πλάι του άλλου, ανεξάρτητα από ε, εθνικότητες, θρησκείες ή τη γεωγραφική διάσταση. Είμαι εδώ λοιπόν στον, ε, στο σπίτι των ευρωπαϊκών λαών. Αυτό το ευρωπαϊκό σπίτι δεν ε, γεννήθηκε σε μια μέρα μόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε μετά από αιώνες πολέμων, μετά από τρομερές αιματοχυσίες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ήταν οι χώροι όπου αποφασίστηκαν πόλεμοι μεταξύ των ε, εθνών της Ευρώπης και ακριβώς μετά την πικρή πείρα του πρώτου και του δεύτερου παγκόσμιου πόλεμου ως πόρισμα από αυτή την πικρή πείρα προέκυψε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από καιρού λοιπόν εις καιρών προκύπτουν δυνάμεις που προσπαθούν να επικρατήσουν επί των ανθρώπων. Το Ισλαμικό κράτος ε, είναι νέο φαινόμενο, αλλά η φύση του δεν είναι καινούρια. Τέτοια φαινόμενα επανεμφωνίζονται με διαφορετικά ονόματα και διαφορετικές μορφές σε όλες τις φάσεις της ιστορίας. Είναι μια βούληση που θέλει να παρεκκλίνουν οι λαοί από την πορεία τους, που επιτίθεται στους ανθρώπους που επιτίθεται και στον άμαχο πληθυσμό, σε γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, είναι ε, μια δύναμη που θέλει να χύσει αίμα. Γι' αυτό πρέπει να αντιδράσουμε όλοι ενιαία και να αντιδράσουμε ακριβώς σε επίπεδο ανάλογο της απειλής. Γιατί μη θεωρείτε ότι το Ισλαμικό κράτος είναι μόνο εχθρός του Ιράκ. Είναι εχθρός ανθρωπότητας. Είναι δικό σας εχθρός όσο και δικός μας. Είναι πρόκληση αντιμετώπιση του για σας όπως και για μας. Και η Ισλαμική πρωτεύουσα προσπαθεί, συγγνώμη, το Ισλαμικό κράτος προσπαθεί ε, να χύσει αίμα και στις δικές σας πρωτεύουσες. Προσπαθεί να σκοτώσει τα δικά σας τα παιδιά όπως σκοτώνει και τα δικά μας. Προσπαθεί να ατιμώσει τις γυναίκες και τις κόρες μας και τις δικές σας να ετοιμάσει συγγνώμη, προσπαθεί να σκοτώσει και να υποδηλώσει παιδιά παντού. Μέσω του αγώνα μας κατά του ΝΤΑΕΣ, του Ισλαμικού κράτους, προσπαθούμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Αυτό είναι ο μόνος δίκαιος πόλεμος. Ο πόλεμος για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όλοι οι άλλοι πόλεμοι είναι απαράδεκτη. Είναι πόλεμη για οικονομικό ή γεωγραφικό όφελος. Αλλά ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας είναι πόλεμος κατά αυτών που θέλουν να δολοφονήσουν την αξιοπρέπεια. Η Μοσούλη είναι η δεύτερη από πλευράς πληθυσμού πόλη του Ιράκ. Αλλά στην πραγματικότητα ο πόλεμος δεν αφορά την Μοσούλη. Αφορά οποιοδήποτε έδαφος όπου εξαπλώνονται αυτές οι δυνάμεις του κακού. Οι δυνάμεις αυτές ε, προσπαθούν να θίξουν το Ιράκ του οποίου ο πολιτισμός έχει 6.000 χρόνια ιστορίας. Η Νασερία, η Μπασόρα, η Βαλαουιά είναι κέντρα του ανθρώπινου πολιτισμού και το ΝΤΑΕΣ προσπαθεί ακριβώς να εξαλείψει αυτόν τον πολιτισμό που έχει 6.000 χρόνια πορεία. Αυτές οι δυνάμεις του κακού που συγκεντρώνονται ε, στη Μοσούλη από σχεδόν όλες τις γωνιές του πλανήτη. Όπως ξέρετε υπάρχουν πάνω από 100 εθνότητες που συμμετέχουν στις δυνάμεις του Νταέσου. Υπάρχουν Αμερικανοί, Αυστραλοί, Καναδοί, Ευρωπαίοι και φυσικά ε, υπήκοοι διαφόρων αραβικών χωρών. Να μην σας εκπλήσει λοιπόν το γεγονός αυτό διότι οι τερροριστικές επιδιώξεις ε, δεν είναι κάτι που προέρχεται και γεννάται μόνο στην περιοχή μας. Παντού υπάρχουν τέτοιες στάσεις. Αυτά τα άτομα ε, μπορεί να είναι υπήκοοι μεγάλων δημοκρατικών λαών, αλλά φυσικά δεν εκπροσωπούν τους λαούς αυτούς, ούτε τα κοινοβούλια, ούτε τις αξίες αυτών των χωρών. Εμείς κρίνουμε τις χώρες σας ε, μέσω των τοποθετήσεων που είναι καθόλου έντιμες των θεσμών σα, των κυβερνήσεών σα, των μη κυβερνητικών οργανώσεών σα που έχουν στηρίξει το Ιράκ κατά τον ΤΑΕΣ. Η σημερινή μάχη λοιπόν δεν αφορά μόνο την Μοσούλη ή ε, την κυβέρνηση του Ιράκ. Είναι ένας ε, πανανθρώπινος αγώνας για την προστασία των πανανθρώπινων ιδανικών. Είναι ένας παγκοσμιοποιημένος πόλεμος κατεξοχήν. Είναι ένας πόλεμος που διεξάγεται παντού στον κόσμο. Αυτό έχουν επιβάλει. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 στη Νέα Υόρκη. Κατόπιν μεταφέρθηκε στη Μαδρίτη, σε άλλα μέρη της Ευρώπης, στην ε, Μέση Ανατολή. Και ο πόλεμος τώρα βλέπουμε ότι έχει εξαπλωθεί και στη Συρία και στο Ιράκ. Είναι ίσως ο πιο σημαντικός πόλεμος ε, που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα έχουν υπάρξει πόλεμοι που κράτησαν περισσότερο και είχαν περισσότερα θύματα, αλλά οι πόλεμοι αυτοί δεν είχαν στο στόχαστρό τους με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο βαθμό τα παιδιά. Δεν είχαν με τέτοιο τρόπο και σε τέτοια ένταση στο στόχαστρό τους να βιάζουν τις γυναίκες και μετά να τις καίνε, όπως έγινε στο Τάλαφάρ με τις γυναίκες των Τουρκομάνων είναι για μας ένας ιερός πόλεμος, γιατί είναι πόλεμος για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όχι μόνο στο Ιράκ. Δεν είναι μόνο θέμα αυτό Προασπίζουμε όλες αυτές τις αξίες. Είναι ένας πόλεμος για κάθε άνθρωπο. Είναι ένας ιερός πόλεμος κατά ενό φαινομένου που είναι στίγμα για τις κοινωνίες μας. Ίσως κρατήσει πολύ γιατί είναι ένας πόλεμος μεταξύ των δυνάμεων του καλού και του κακού. Είναι ένας πόλεμος του πολιτισμού και των αξιών κατά των δυνάμεων του κακού και της επιθετικότητας του κακού. Ίσως να μας κοστίσει πολύ αυτός ο πόλεμος. Οπωσδήποτε θα κοστίσει. Και ο πληθυσμός του Ιράκ σήμερα ε, πληρώνουν το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του τιμήματος. Χύνουν το αίμα τους, καταστρέφονται οι υπηρεσίες τους, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να το πληρώσουμε. Το Ιράκ είναι μια πλούσια χώρα, έχει διάφορους πόρους. Πρώτα απ' όλα έχουμε το πετρέλαιο. Επιπλέον είμαστε η χώρα της Μεσοποταμία, του Τίγρη, του Εφράτη, της Γεωργίας, του τουρισμού. Είμαστε μια πλούσια χώρα σε πρώτες ύλε και ορυκτά. Αλλά σήμερα είμαστε σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Η τιμή του πετρελαίου, όπως ξέρετε, έχει πέσει πάρα πολύ. Και το κόστος ε, των στρατιωτικών μας δαπανών μας έχει οδηγήσει σε πολύ σοβαρό έλλειμμα του προϋπολογισμού μας. Και θέλω να ευχαριστήσω όλες τις κυβερνήσεις που στήριξαν το Ιράκ μέσω οικονομικής βοήθειας. Το Ιράκ δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτούς που το στήριξαν ιδίω στη δύσκολη φάση που περνάει τώρα. Όπως είπε και ο φίλος μου ο πρόεδρος, Παρόμοιες τέτοιες καταστάσεις έχουν προκύψει και άλλες φορές στον κόσμο. Πρέπει όμως ακριβώς να βγάλουμε διδάγματα από το παρελθόν. Και το δίδαγμα, και το δίδαγμα πρέπει να είναι ότι πρέπει από κοινού να το αντιμετωπίσουμε τον ΤΑΕΣ, γιατί αν δεν το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί θα προκύψει και σε άλλα μέρη του κόσμου. Το ΤΑΕΣ στρέφεται κατά όλων των λαών, κατά των παιδιών, κατά των γυναικών, κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι τιμή για μας που είμαστε στην πρωτοπορία της καταπολέμησης αυτών των εχθρών της ε, ανθρωπότητας και του πολιτισμού. Υποθέτω ότι θέλετε να μάθετε τι γίνεται στη Μοσούλη. Είναι μια πόλη στο βορρά της χώρας μου, η δεύτερη σε πληθυσμό μετά από τη Βαγδάτη. Εγώ για παράδειγμα φίτησα και έχω πτυχίο ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Μοσούλης. Άρα γνωρίζω πολύ καλά τους κατοίκους ε, της πόλης αυτής. Έζησα σε αυτή την πόλη τόσα, τόσα χρόνια και γνωρίζω καλά αυτή την πόλη. Είναι μια πόλη που είναι περίφημη για το επίπεδο του πανεπιστημίου της και ιδιαίτερα για τους γιατρούς της, για τους αξιωματικούς του στρατού, προέρχονται από τη Μοσούλη και είναι και σημαντικό οικονομικό κέντρο το οποίο κατελήφθη από τους τρομοκράτες αξιοποιώντας ε, κάποιες διχόνες που υπήρχαν στην ε, πόλη αυτή και τη στήριξη κάποιων άλλων χωρών. Αλλά η αντίσταση των κατοίκων της πόλης, η αντίσταση αυτή που προκάλεσε μαζικές εκτελέσεις, ήταν ε, πραγματική και παρά τα βάσανά της η πόλη αυτή έμεινε όρθια και ήρθε η ώρα να απελευθερωθεί η Μοσούλη να ξαναγίνει τμήμα της χώρας της να ξαναγίνει τμήμα του Ιράκ και τμήμα της ελεύθερης ανθρωπότητας οι κάτοικοι της Μοσούλης έχουν διαφορετικές θρησκείες και διαφορετικές εθνικές προελεύσεις είναι ένα μείγμα και Έχουμε λοιπόν ε, καταρτήσει το σχέδιο της επιχείρησης για να καταλάβουμε την πόλη, για να ληφθεί βοήθεια, να αποσταλεί βοήθεια, να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες που πιθανώς θα προκύψουν και για να μπορέσουμε να οργανώσουμε τις αναγκαίες υπηρεσίες, ιδιαίτερα τις ιατρικές υπηρεσίες. Τα έχουμε προετοιμάσει όλα αυτά σε συνεργασία με τους συμμάχους μας, ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους, τους Αυστραλούς, αλλά και τους Αμερικανούς από το βήμα αυτό. στρέφομαι λοιπόν προς όλους εσάς για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας προς όλους τους φίλους και τονίζω ότι όταν θα νικήσουμε, θα νικήσουμε για όλη την ανθρωπότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πραγματικά για τη δυνατότητα αυτή. Σας ευχαριστώ για αυτή την τοποθέτησή σας. Να σας πω ότι έχουμε έξι συναδέλφους, εφτά. Ζήτησαν το λόγο. 8 8 συναδέλφους λοιπόν επειδή έχουμε μισή ώρα θα ήθελα να μιλήσει ο καθένας για δύο λεπτά και μετά να επιτρέψουμε στον κύριο Υπουργό να απαντήσει. Να Ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Αντάκτουσον. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο αυτό στις αρχές ε, Φεβρουαρίου φέτος ε, πέρασε ένα ψήφισμα για την κατάσταση στο Ιράκ ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τι μειονότητε. Αυτό το ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η μεγαλύτερη ομάδα στο Κοινοβούλιο, στην οποία ανήκω και εγώ και εκεί πέρα. Αναφερθήκαμε στις ε, ακρότητες ε, που υφίστανται αυτές οι μειονότητες ε, ως γενοκτονία που διαπράττει το Ισλαμικό κράτος. Ε, έχοντας αυτό βάση θα ήθελα να θέσω το ζήτημα των αυτοχθόνων αυτών μειονοτήτων και την κατάσταση η οποία θα προκύψει μετά την απελευθέρωση της Μουσούλης. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Τι χρειάζεται έτσι ώστε χριστιανοί, σιροχαλδαίοι Γεζίδιδες ε, και Τουρκομάνοι να μπορέσουν να επιστρέψουν στις ε, περιοχές από όπου καλαγόνται στην Νινεβή, Σινιάρ και τα Λαφάτα. Νομίζω πως είναι κρίσιμο το ερώτημα και γνωρίζω τις προκλήσεις και τα προβλήματα αλλά θα ήθελα να ακούσω την δική σας ε, την άποψη. για το τι θα γίνει μετά την απελευθέρωση της ε, Μοσούλης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Χάν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Σαλαμαλέκομ και καλώς ήρθατε. Και σας συγχαίρω για το χθεσινό Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιρακ και Νομίζω πως ε, αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μοσούλη κατά του Ισλαμικού κράτους ελπίζω να, οι επιχειρήσεις να τελειώσουν ε, σύντομα και να είναι επιτυχής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είναι η ανησυχία για τον ανθρωπιστικό αντίκτυπο της επίθεσης. Ειδικά το τι θα σημάνει αυτό για τους πρόσφυγες και τι έχει κάνει η κυβέρνησή σας ήδη για να το αντιμετωπίσει. Αντιλαμβάνομαι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποσχεθεί 95 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει. Πώς θα σίγουρευτείτε ότι θα φτάσουν αυτά τα κονδύλια στους ανθρώπους ε, για τους οποίους προορίζονται και κάτι άλλο το οποίο αναφέρθηκε ο συνάδελφος τα ζητήματα των μειονοτήτων. Να σας ρωτήσω το εξής. Όλο αυτό το σενάριο του ΝΤΕΣ ε, και το τι συμβαίνει το τι συνέβη στην Μοσούλη σχετιζόταν ε, και βεβαίως με τον σεχταρισμό, την αντιπαλότητα μεταξύ των κοινοτήτων. Τι βήματα έχουμε γίνει λοιπόν για να μην ξαναπέσουμε σε αυτή την κατάσταση έτσι οι διάφορες κοινότητες, μειονότητες και πλειονότητες να θεωρούν ότι είναι μέρος του Ιράκ. Και τέλος, ανέφερα το ε, Ερμπίλ ε, το επισκέφθηκα. Έχω δει την κατάσταση και τις προσπάθειες ε, της κουρδικής κυβέρνησης με τους πρόσφυγες. Ένα ζήτημα εκεί ήταν κάποιες διαφωνίες στα οικονομικά με την ε, κεντρική κυβέρνηση. Έχει υπάρξει κάποια βελτίωση από αυτό. Ευχαριστώ. ως Κόζο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Δεν θα χρειαστώ δύο λεπτά. Πρώτον, συμφωνώ με αυτό που είπαν κάποιοι συνάδελφοι για τις ε, στρατικές δυνάμεις που απελευθερώνουν το Μοσούλ. Ε, θα αποφύγουν τα λάθη που έγιναν ε, κατά ορισμένων μενοτήτων το 2011. Δεύτερον, για την επίτευξη των στόχων για, από τις αεροπορικές επιθέσεις δεν ε, έχουμε τις πληροφορίες που θα θέλαμε. Και κάτι που διάβασα στην Ισπανική, στον Ισπανικό τύπο. Οι δυνάμεις που επιτίθεται θα ανοίξουν διάδρομο για να πάνε στις διπλανές χώρες ε, οι μαχητές του Νταέσ. Αν είναι αλήθεια αυτό θα ήταν σκανδαλώδες. Δύο λεπτά κυρία Λόχ Μπίλερ. Ναι, ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε για να συζητήσετε μαζί μας και ευχαριστώ και για τις δηλώσεις σας. Έχω δύο ερωτήσεις. Το ένα αφορά τον τρόπο διεξαγωγής της ε, μάχης και πώς βλέπετε την απελευθέρωση της Μοσούλης. Ε, το Σεπτέμβριο όταν απελευθερώθηκε η Φαλούτζα υπήρχαν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μαζικές ε, ομαδικές εκτελέσεις κτλ και η κυβέρνηση του Ιράκ είπε ότι θα το ερευνήσει και, και θα προχωρήσει μέτρα και βεβαίως στην απελευθέρωση της ε, Μοσούλης είπατε ότι ειδικά κάποια, κάποιες ηθικές ένοπλες ομάδες ε, δεν θα είναι μέρος της προσπάθειας τώρα από το Ρέι στο Reuters διάβαζα πως ε, κάποιες σιητικές δυνάμεις ε, πολεμούν στο πλευρό του Ιρακίνου στρατού. Ειδικά σε μια κοιλάδα στα δυτικά της ε, πόλης. Το θέμα δεν είναι... Το θέμα είναι ότι βεβαίως πλήττονται και πάρα πολύ άμαχοι, όχι μόνο οι μαχητές του Ισλαμικού κράτους από αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ κύριο Καστάλτο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, εξοχότητε. Σαλαμαλέκουμα. Ε, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Παρακολουθούμε τις προσπάθειες ε, που καταβάλλονται μαζί και με τους Πέσμεργα. Ε, εγώ θέλω να σας μιλήσω για τα όσα ακούμε από την Τουρκία. Φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες εντάσεις ανάμεσα στην Ιρακινή κυβέρνηση που εσείς εκπροσωπείτε και την τουρκική και συγκεκριμένα για τη συμμετοχή τουρκικών δυνάμεων στην μάχη για την απελευθέρωση της Μοσούλης. Ε, Μάλιστα πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράκ και φαίνεται ότι υπάρχει και μεγάλη κοινότητα τουρκομάνων, δηλαδή κοντινή στι θέσει τη τουρκική κυβέρνηση. Ε, μάλιστα εκφράστηκαν και θέσει όπω αυτή τη παραστατική οργάνωση Al-Sad Al-Shabi που λέει ότι θεωρεί την τουρκική ε, δύναμη εξωτερική ξένη δύναμη εχθρική και είναι έτοιμη να του ε, πυροβολήσουν, να του συναντήσουν. Επίσης υπάρχει διεθνής δύναμη στη ε, Ερμπίλ, στην Ερμπίλ που μπορεί να κινηθεί και να ληφθεί στην περιοχή. Τώρα, δεδομένου ότι είναι πολύ έντονες αυτές οι ε, δηλώσεις και ακατάλληλες από πλευρά του Προέδρου Ερντογάν κατά του Πρωθυπουργού Χαϊδέρα Λαμπάντη, εσείς τι γνώμη έχετε, πιστεύετε πως ε, θα μπορέσει να υπάρξει κάποια συμφωνία με τις ε, περιφερειακές ε, αρχές των Κούρδων και τι πιστεύετε θα γίνει μετά την απελευθέρωση της πόλης. Δεύτερη μου ερώτηση αφορά τη γνώμη σας για την κατάσταση στη Συρία, όπου υπάρχουν και οι παραστατικές, παραστατικές ε, ομάδες, όπως η Αλφάτ και άλλοι παραστατικές οργανώσεις ε, Ιρακινής προέλευσης που συμβάλλουν στο να μετατρέπεται αυτή η μάχη, η σύγκρουση σε ανοιχτή σύγκρουση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ποια είναι η προοπτική της Ιρακινής κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποργκέτσιο, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και ε, ε, χαιρετίζω και ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό που μας τιμά με την παρουσία της. Εγώ συνδέομαι με τα όσα είπε ο κύριος Καστάλτο για την Τουρκία, γιατί διαβάζω ότι ο πρόεδρο Ερντογάν έκανε μια δήλωση σύμφωνα με την οποία ε, η Τουρκία και οι Ηνωμένε Πολιτείε συζητούν την υπόθεση μιας κοινή ε, στρατιωτικής επιχείρησης για να μπορέσουν να εκδιώξουν το ίσις από το χειρό, της, ε, το χειρό του στη Συρία, την Ράκα αυτά εντό εισαγωγικών. Και άλλο ένα, άλλη μια είδηση που φαίνεται να είναι πολύ σοβαρή υπό το φως ε, των κινδύνων για τον άμαχο πληθυσμό είναι το γεγονός ότι το ίσις, ε, το ΝΤΑΕΣ μπορεί αυτή τη στιγμή λέει να χρησιμοποιήσει και χημικά όπλα γιατί φαίνεται ότι, υπάρχει, ότι έχει στην κατοχή του διάφορα χημικά όπως ε, χλώριο και άλλα. Και έπειτα τι θα γίνει με αυτούς τους ξένους μαχητές. Θα φύγουν προς τη Συρία. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι μυστικά έχουν γίνει διαπραγματεύσεις ε, για να υπάρξει μία ασφαλής έξοδος τους. Αλλά πού θα πάνε, θα πάνε και αυτοί στη Συρία και έπειτα ο Αλμπαγκδάτη αφού ξέφυγε από την έφοδο είναι ακόμα εκεί στην Μοσούλη ή έχει μετακινηθεί κάπου πιο σε μεγαλύτερη ασφάλεια στη Συρία. Ε, υπάρχει, έχουν ε, ψήγματα αλήθεια στα όσα καλούν τον πληθυσμό σε λαϊκή εξέγερση. Μπορεί δηλαδή να περιμένουμε από πλευράς των πολιτών να στηρίξουν αυτή την ιδέα της απελευθέρωσης με τέτοιο τρόπο. Τέλος, ποια είναι η δική σας γνώμη για τους κινδύνους που μπορεί να διατρέχει το Ιταλικό τάγμα που συμμετέχει στην μάχη της Μοσούλης γιατί είναι μια συνήθιστη επίθεση και μπορεί να είναι μια από αυτές τις επιχειρήσεις προπαγάνδας όπου δυστυχώς το ίσις έχει δείξει ότι είναι πολύ ικανό. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη για τις πολυάριθμες ερωτήσεις. Ο κύριος Επιτίδιος, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε εξοχότατε. Έχω τρεις ερωτήσεις για σας. Η πρώτη ερώτηση ε, είναι η εξής έχει δώσει η Ιρακινή κυβέρνηση στι ένοπλε δυνάμει που διεξαγάγουν τι επιχειρήσει οδηγίε, ούτω ώστε να περιορίσουν τι απώλειε ε, των αμάχων. Μια και γνωρίζετε τη Μοσούλη, γνωρίζετε αν υπάρχουν καταφύγια στο οποίο μπορεί να καταφύγει ο πληθυσμό εκεί ή θα χρησιμοποιηθεί ω ε, ανθρώπινη ασπίδα από τι δυνάμει του ΆΙΣΙ. Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξή. Ε, μία από τι δυνάμει που είναι σύμμαχο του Ιρακινού στρατού είναι η παραστρατιωτική οργάνωση Ασάντα Αλ Σάμπι ή Popular Mobilization Forces, όπως ε, λέγονται. Αυτοί είναι Σιήτες. Ε, έχει ληφθεί κάποια πρόνοια από την Ιρακινή κυβέρνηση, ώστε να μην ε, προβούν σε βιοπραγίες εναντίον του πληθυσμού της Μοσούλης που στην πλειοψηφία του είναι Σουνίτες. Και τρίτο, πώς σχολιάζεται την εμπλοκή της Τουρκίας στην όλη ε, διαμάχη, στον πόλεμο αυτόν. Πρόσφατα ο πρόεδρος Ερντογκάν είπε ότι το Ιράκ είναι μια γη τουρκική. Τι, περιμένετε, τι προσδοκάτε από την εμπλοκή της, από Τουρκίας σε αυτή τη ε, μάχη ή τι φοβάστε από αυτή. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, now... Ευχαριστώ. Η κυρία Κάτι Πύρη. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εφόσον τώρα αρχίζει η απελευθέρωση της Μοσούλης, ε, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους Ανδρίους των Ιρακινών Δυνάμεων και των Πεσμέργα. Η ερώτηση του συνάδελφου Καστάλτο αφορά την πρόσφατη ένταση μεταξύ Βαγδάτης και Άγκυρας και οι τελευταίες πληροφορίες ότι η τουρκική αεροπορία συμμετείχε στις αεροπορικές επιθέσεις κατά της Μοσούλης. Θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η άποψή σα επ' αυτού. Ακούσαμε ότι τώρα, που είναι τρίτη μέρα της επίθεση, χιλιάδε Ιρακινοί διαφεύγουν στη Συρία. 5.000 έφτασαν στο στρατόπεδο Αλ-Χοκ στη Συρία και ορισμένοι και χιλιάδε άλλοι είναι μπλοκαρισμένοι στα σύνορα. Και η μη κυβερνητική οργάνωση, οργάνωση Σώστε τα Παιδιά έβγαλε μια δήλωση που λέει ότι οι συνθήκε ε, είναι από τι χειρότερε που έχουν δει ποτέ και περιμένουν και πολλέ άλλε χιλιάδε να φτάσουν σύντομα. Μπορείτε να μας πείτε εάν υπάρχουν επίγοντα προγράμματα για να βοηθηθούν οι άμαχοι που προσπαθούν να διαφύγουν από την Μοσούλιο. Κύριος Φανμπάλεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι τιμή μας η παρουσία σας, κύριε Υπουργέ. Να σας ρωτήσω. Οι Ρώσοι συμμετέχουν στην περιοχή Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, η Τουρκία και πολλοί άλλοι. Ο στόχος είναι η εξάλληψη του Ισλαμικού κράτους και, των εδαφών, και να, η απελευθέρωση των εδαφών που κατέχει. Πώς βλέπετε τη συνεργασία μεταξύ όλων αυτών ορισμένοι, όχι μόνο δεν συνεργάζονται, αλλά ε, ο ένας πολεμάει τον άλλον. Πώς τα βλέπετε αυτά. Ευχαριστώ η κυρία Γκόμες. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Και εγώ είχα πάει πέρσι στο Ερμπίλ. Είδα εκεί τους Πεσμεργά που ετοιμαζόταν να πάνε στη Μοσούλη, αλλά ήθελαν στήριξη από τις σουνητικές δυνάμεις γιατί ε, ήθελαν να αποφύγουν τα αντίπεινα και κατηγορίες περί ρεβανσισμού. Πρόκειται για έναν ευρύτερο συνασπισμό και θα διατηρηθεί και ο Ιρακινός στρατός θα ξεπεράσει τις αιτίες Ε, οι οποίες οδήγησαν στην πτώση της ε, Μοσούλης. Λοιπόν, για τον ρόλο της Τουρκίας μπορείτε να μας πείτε ε, τι άποψη έχετε για το ότι ενισχύει το ΝΤΑΕΣ η Τουρκία και του δίνει τη δυνατότητα να επιχειρεί στη Συρία και στο Ιράκ. Τώρα θεωρείτε ότι στόχος τους είναι να περιορίσουν τους Κούρδους ή έχουν πραγματικά εδαφικές και υδάτινες φιλοδοξίες ε, εις βάρος του Ιράκ και της Συρίας και τι ε, περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να σας ε, βοηθήσει να ξαναχτίσετε τις περιοχές στις οποίες μπορούν να επιστρέψουν οι μειονότητες και οι πρόσφυγες, Σιντζάρ, Νινεβή κτλ. Σας ευχαριστώ κύριε Λίτς. Α, ναι, Λίτς, λέγομαι Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σε αυτά τα οποία προσέθεσε η κυρία, είπε η κυρία Γκόμες. Τι θα κάνετε με τα όσα έγιναν στην χώρα, ειδικά όσον αφορά τη μεταβατική δικαιοσύνη, θα υπάρξει μια διαδικασία συμφιλίωσης. Αναφέρθηκε σωστά και το ζήτημα του Ισλαμικού κράτους και του υπόβαθρου που υπάρχει. Και βεβαίω ε, τι θα κάνουμε με την Συρία και τι δυνάμει που εμπλέκονται εκεί και πώ θα υπάρξει δικαιοσύνη διεθνώ. Δηλαδή το Ιράκ ε, έχει, είναι ήδη συμβαλόμενο μέρο στο διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Και θα πρέπει νομίζω να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Βλέπουμε τόσα πράγματα στην περιοχή και πρέπει το θέμα αυτό να το προωθήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ε, ασχολείται με το ζήτημα αυτό και αναρωτιέμαι πώς ε, το βλέπετε και στην, ε, στο ευρύτερο πλαίσιο αλλά και όσον αφορά την ε, κατάσταση στο εσωτερικό του Ιράκ. Σας ευχαριστώ και εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά στη χώρα σας. Σας ευχαριστώ. Κάνατε αρκετές ερωτήσεις που κάλυψαν πολλές πτυχές που αφορούν ιδιαίτερα τη Μοσούλη, αλλά έγιναν και ερωτήσεις ε, πολλές παρόμοιες, ε, όπως αυτές που αφορούσαν την Τουρκία. Λοιπόν, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ναι, Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Δέκα ομιλητές ε, έθεσαν ερωτήσεις που στην ουσία καλύπτουν όλες τις πτυχές της κατάστασης. Για να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις ε, θα έπρεπε να έχω στη διάθεσή μου πολύ χρόνο. Επιτρέψτε μου ωστόσο να είμαι σύντομος ε, και περιεκτικός και θα ζητήσω τη βοήθεια των διερμηνέων, λέει ο Υπουργός. Όσον αφορά την κατάσταση που ισχύει στο Ιράκ για τις μειονότητες, τις αποκαλούμε μειονότητες, δεχόμαστε αυτή την έννοια, αυτή την ιδέα, αλλά δεν υπάρχει, δεν, δεν πρόκειται για μειονότητες ε, αυτό καθ' αυτό, γιατί είναι σημαντικές για το Ιράκ. Είναι αριθμητικά μικρότερες ομάδες, αλλά η εργασία, ο πολιτισμός, η κληρονομιά που έχουν αφήσει στη χώρα μας δεν αποτελούν για αυτές ε, αχίλιοπτέρνα. Αντιθέτως, πρόκειται για μία δύναμη. Είναι ναι αλλά έχουν παίξει πολύ ε, μεγάλο ρόλο για τον οποίο είμαστε περήφανοι. Μάλιστα, αντιπροσωπεύονται στις ένοπλες δυνάμεις μας. Έχουμε, δηλαδή, έχουμε ε, χριστιανούς, ε, γιασίδι στις ένοπλες δυνάμεις μας, οι ε, χώροι λατρείας, όπως ο Άγιος Σώστης, η Εκκλησία του Άγιου Σώστη, έπεσε θύμα βομβαρδισμών όπως το ίδιο έγινε και με τζαμιά στη χώρα μας. Ε, υπάρχουν εκπρόσωποι δε των μειονοτήτων στην κυβέρνηση, στον διοικητικό μας μηχανισμό, σε όλα τα επίπεδα και όλο το πληθυσμιακό, μοσαϊκό, εθνοτικό και θρησκευτικό αντιπροσωπεύεται στις κρατικούς μας θεσμούς και οι θυσίες ε, δεν ήταν λίγες. Ξέρετε τι έχει γίνει με τους Γιαζίδη στην πόλη Σινζάρ, που τα κορίτσια ε, βιάστηκαν, τα παιδιά απολύθηκαν στη Συρία. Όταν λέμε Ιρακινός λαός, εμείς δεν ε, κάνουμε διακρίσεις ανάμεσα στι μειονότητες, γιατί όλες αυτές οι μειονότητες υπερασπίζουν τη χώρα τους και σχηματίζουν κοινό μέτωπο απέναντι στον εχθρό. Δεν μιλάμε λοιπόν για μειονότητες, πρόκειται για ένα πολιτιστικό και ε, πολιτιστικό φαινόμενο το οποίο υπάρχει στο Ιράκ ανέκαθεν. Από την απαρχή της ανθρωπότητας. Ξέρετε την στήλη του Αμυραμπή, το 1572 ήδη μιλούσε, ανέφερε τα ανθρώπινα δικαιώματα. 3.000 περίπου χρόνια πριν από τον Ιησού Χριστό. Μιλούσε για ανθρώπινα δικαιώματα και για δικαιώματα της γυναίκας. Ο Ιρακινός πολιτισμός οδηγεί στο ότι οι διάφορες συνιστώσεις αυτού του Ιρακινού μοσαϊκού να έχουν πάντοτε ζήσει μεταξύ τους ειρηνικά. Οι Ιρακινοί ποτέ ε, δεν ρωτάνε ποιος είναι χριστιανός, ποιος είναι γιασίτη. Όλες οι εθνότητες είναι στόχος, γιατί τον Ταΐς τα έχει βάλει με όλους δεν είναι ο πόλεμος θρησκευτικός. Είναι πόλεμος κατά της ανθρωπότητας και κατά του λαού του Ιράκ, των πολιτών, των ειρηνικών πολιτών του Ιράκ. Είναι πραγματικά ένας πόλεμος ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Δυνάμεις του κακού, στους οποίους πολλούνται όπλα. Το ίδιο και για τους Τουρκμένους, που, Τουρκμένους που είναι μεγάλη συνιστόσα του κοινωνικού και θρησκευτικού ιστού του Ιράκ έχουν προσφέρει πολλά, έχουν ε, θυσιαστεί και υπό το παλιό καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν. Όλα τα παιδιά του Ιράκ, όποια και αν είναι η θρησκεία τους, συμβάλλουν στην οικοδόμηση του αυριανού Ιράκ. Σας ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήρια και για τις ευχαριστίες σας, αλλά θέλω να επιμείνω στο γεγονός ότι... Οι ανθρωπιστικές προσπάθειες είναι σημαντικές. Προσπαθήσαμε να μειώσουμε τον αριθμό των εκτοπισμένων πριν την ε, προαναγγελθήσα μάχη, γιατί δεν πρόκειται μόνο για την απελευθέρωση της ε, Μοσούλης. Ε, φυσικά ετοιμάσαμε την μάχη. Είμαστε τώρα στην μάχη, στη φάση της μάχης και μετά θα πρέπει να περάσουμε στην τρίτη φάση γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων της Μοσούλης στα σπίτια τους. Είναι μια μεγάλη πόλη Πολλά εκατομμύρια κόσμος κατοικεί εκεί και θέλουν να μπορούν να έχουν υπηρεσίες ε, νοσοκομιακή περίθαλψη για τους ίδιους και τα οικογένειέ τους. Η προετοιμασία της μάχης συμβαδίζει με την προετοιμασία παροχής υπηρεσιών κοινωνικών αλλά και υγειονομικών σε αυτή τη τόσο δύσκολη ε, κατάσταση. Όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη στην προσπάθεια προετοιμασίας θα προσπαθήσουμε να φροντίσουμε από ανθρωπιστικής άποψης όσο γίνεται περισσότερο τον ε, άμαχο πληθυσμό και τα κονδύλια που έχουν δοθεί, έχουν προσφερθεί στο Ιράκ έχουν ξεπεράσει τα 2 δις δολάρια. η ΕΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο προσέφεραν 100 εκατομμύρια την περασμένη εβδομάδα και δεν ξεχνάμε φυσικά την Ευρωπαϊκή Ένωση που προσέφερε επίσης άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ και όλα αυτά βεβαίως θα ληφθούν υπόψη. Οι δωρητές μας μπορούν να είναι ήσυχοι διότι τα κονδύλια αυτά δαπανώνται σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Όποια και αν είναι η εθνοτική θρησκευτική ε, προτίμηση του καθενός, και θυμάμαι το δεύτερο μισό του δεκαετία του 60, γύρω στο 1966, είδαμε την καλή, την αγαστή συνύπαρξη ανάμεσα στις διάφορες ε, ε, συνιστώσεις της πόλης της Μοσούλης ε, φάνηκε το Νταές και φάνηκε να υπερασπίζει τους Σουνίτες ενώ οι Σουνίτες δεν είχαν ζητήσει κάτι τέτοιο και το πρόσχημα του ΑΕΣ ήταν ότι υποστήριζαν τους Σουνίτες. Γι' αυτό υποτίθεται ότι κατέλαβαν αυτή την πόλη. Πρόκειται για ψέματα, για ψευδείς φήμες. Όσον αφορά τις αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και τις περιφερειακές κυβερνήσεις, αυτές ανήκουν στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή η κεντρική κυβέρνηση, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ε, ε, συνεργάζεται αρμονικά με τις επαρχίες. Είναι το θέμα του πετρελαίου και της ε, κατανομής του που δεν είχε ρυθμιστεί. Η κυβέρνηση μπόρεσε να μειώσει ε, να περιορίσει μάλλον αυτή την ανταπεράθεση. Τώρα όσον αφορά την σύσταση των ε, Ιρακινών ε, ενόπλων δυνάμεων. Το Υπουργείο Αμήνης έχει συγκεντρώσει εθελοντές, αλλά έχει γίνει και η στρατολόγηση των εφέδρων Ακόμα και ε, το, ο, Σερ ε, ζήτησε να ξεχάσουμε, να βάλουμε κατά μέρος τι σκεφτικές μας διαμάχες ώστε να μπορέσουν όλοι να λάβουν μέρος στην μάχη για την αξιοπρέπεια της χώρας. Οι ενόπλες δυνάμεις αντιπροσωπεύονται από το Πρωθυπουργό και το Ιρακινό Σύνταγμα δίνει στον Πρωθυπουργό δύο σημαντικά καθήκοντα. Πρώτον, την Προεδρία του, Συμβουλίου, του Υπουργικού Συμβουλίου και στη συνέχεια την αρχηγία των ενόπλων δυνάμεων. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν έχει αυτές τις δύο αρμοδιότητες. Θέλω να αποφύγουμε τις ε, θρησκευτικές διενέξεις μεταξύ των διαφόρων ε, θρησκειών στη χώρα μας. Θα το λέω πολύ ειλικρινά. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή θρησκευτικές διενέξεις μεταξύ των διαφόρων τμήματων της ε, Ιρακινής κοινωνίας. Ο λαός του Ιράκ είναι ένας μικρόκοσμος ε, διαφόρων ε, κοινωνιών. Έχουμε Άραβες, ε, Σουνίτες, Σίτες, Τουρκμένους, Γεζίντι, αλλά δεν ζουν σε γκέτο. Όλες αυτές οι συνιστώσεις συμβιούν σε όλες τις πόλεις και επαρχίες του Ιράκ. Όλες οι περιοχές του Ιράκ έχουν εκπροσώπηση όλων των κοινοτήτων, όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων. Ε, μην πιστεύετε ορισμένες φήμες που διαδίδονται μέσω των ΜΜΕ. Οι Ιρακινοί ζουν σε αγαστή συνεννόηση και σε ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων. Και αυτή η παράδοση ειρηνικής συμβίωσης ε, περνάει από μία γενιά στην άλλη. Εγώ προέρχομαι από την Καρμπάλα που είναι ένας από τους ιερούς τόπους, μάλιστα πιο σημαντικό. Το Βατικανό του Σιητισμού θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Άρα μην πέφτετε σε καμία παγίδα. Μην ακούτε τις ψευδολογίες. Γιατί πολλά λέγονται τα οποία είναι εντελώς αβάσιμα. Δεν πρέπει να τα πιστεύετε. Τώρα, Προετοιμάσαμε αυτήν την ε, επίθεση ε, με πολύ προσοχή και μας πήρε πολύ χρόνο. Γιατί στόχος μας ήταν να μειωθούν στο απόλυτα απαραίτητο οι απώλειες μεταξύ, του ε, μεταξύ των αμάχων. δεν θέλουμε να υπάρξουν διενέξεις μεταξύ Σουνιτών και Σιητών, διότι και οι Σουνίτες και οι Σιήτες, όπως σας είπα, συμβιούν ειρηνικά και αρμονικά μαζί με τους χριστιανούς, τους χαλδαίους και τους γιαζίντι. Πρέπει να ξέρετε ότι μεταξύ των πρώτων ε, μαρτύρων των ε, λαϊκών πολιτοφυλακών, των εθελοντών που στρατολογήσαμε δηλαδή, ήταν Σουνίτες. Αυτές οι στρατιωτικές ε, δυνάμεις, αυτές οι πολιτοφυλακές που δημιουργήσαμε, είναι ανοιχτές για όλες τις κοινότητες εθνοτικές ή θρησκευτικέ. Στη Φαλουζά, για παράδειγμα, θέλω να σας πω το εξή. Δεν είναι σωστοί οι ισχυρισμοί που πολλές φορές βγαίνουν κατά τη διάρκεια της μάχης. Γιατί μπορούν να προκύψουν διάφορες φήμες που είναι εντελώ αδύνατο να ελεγχθούν δεν είναι δυνατόν ε, μια συγκεκριμένη θρησκεία, μια συγκεκριμένη ομάδα να χαρακτηρίζεται άσχημα λόγω κάποιων κακών πράξεων ή της ανικανότητας ενός ατόμου. Τα άτομα μπορεί να κάνουν λάθη, αλλά οι ιδέες και οι κοινωνίες δεν ε, αλλάζουν. Εάν η κυβέρνησή μας έκανε έρευνες, βεβαίως και κάναμε έρευνες για να δούμε εάν υπήρξαν ακρότητες και επιβλήθησαν κυρώσεις σε όσους ε, διέπραξαν εγκλήματα. Με ρωτήσατε εάν ε, οι ε, ε, δυνάμεις θα συμμετάσχουν στην απελευθέρωση της Μοσούλης. Δεν έχουμε σιητικές δυνάμεις. Έχουμε στρατιωτικές μονάδες του Ιρακινού στρατού αυτές θα συμμετάσχουν. Η Πεσμεργά βεβαίω είναι στην περιοχή, γιατί πάντα ήταν εκεί, συμμετέχουν μαζί με τις δυνάμεις λαϊκή κινητοποίηση, όπως αποκαλούμε αυτές τις δυνάμεις, συμμετέχουν μαζί με όλες τις φυλές στην υπεράσπιση του Ιράκ. Έχουμε κάνει κατανομή ρόλων με εγκάρδια συνεννόηση, όσον αφορά τι εντάσει μεταξύ Τουρκία και Ιράκ. Το Ιράκ πάντα σεβόταν την Τουρκία και δεν έχει βλέψεις κατά της Τουρκίας. Όταν για παράδειγμα έγινε το πραξικόπημα στην Τουρκία ήμουν ο πρώτος που ήρθα σε επαφή με την ε, τουρκική κυβέρνηση για να τους εκφράσω την αλληλεγγύη και τη στήριξη προς την τουρκική δημοκρατία. Η απόπειρα πραξικόπηματος δηλαδή. Εάν αλλάξει η κυβέρνηση στην Τουρκία ή αν κάποιοι θέλουν να αλλάξουν την κυβέρνηση με δημοκρατικό τρόπο θα σεβαστούμε το αποτέλεσμα αυτό. Αλλά δεν θα σεβαστούμε ποτέ, δεν θα αποδεικνύουμε ποτέ ένα πραξικόπημα. Και πάντα θα επιλέγουμε ειρηνικέ λύσεις. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία από τις γειτονικέ μας χώρες να παραβιάσει την κυριαρχία του Ιράκ. Είτε είναι το Ιράν, είτε η Σορική Αραβία, είτε το Κουβέιτ, τη Συρία, η Τουρκία, όλες οι... και η Ιορδανία με όλες τις χώρες ε, που συνορεύουμε με τη δική μας έχουμε πολύ καλές σχέσεις αλλά δεν θα αποδεχτούμε ποτέ παραβίαση ή παρέμβαση. Έχουμε συμβούλους και Ευρωπαίους και Αμερικανούς και από άλλες χώρες και από τι γειτονικέ χώρες που συμμετέχουν ως σύμβουλοι. Έρχονται, παίρνουν θεώρηση από το Υπουργείο Εξωτερικών τη χωρα μου, μπαίνουν στην, ε, στο Ιράκ και παραμένουν όσο τους επιτρέπει η βίζα τους. Άρα αυτοί δεν προσβάλλουν την κυριαρχία μας και έχουμε και Ιρανούς και άλλους συμβούλους. Και οι Τουρκομάνοι είναι τμήμα του κοινωνικού μας ιστού. Εκπροσωπούνται και στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση και συμμετέχουν στη μάχη μας. Επεκρίθη ο Αμπάντη από ορισμένου ή από ορισμένε άλλες κοινότητες και εκφράζουμε τη λύπη μας γι' αυτό, αλλά δεν έχουμε το χρόνο, δεν έχουμε την δυνατότητα αυτή τη στιγμή να απαντήσουμε σε αυτές τις επικρίσεις και ιδιαίτερα τις επικρίσεις του Προέδρου Ερντοάν. Εμείς προσλέπουμε σε πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία στο μέλλον. Και πάντα θα θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Η τρομοκρατία είναι απειλή για όλες μας τις χώρες. Αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν την Συρία θα θέλουν να αποσταθεροποιήσουν και να καταστρέψουν και το Ιράκ. Αν αποτύχουμε λοιπόν στο Ιράκ θα αποτύχουμε και στη Συρία. Ορισμένοι ρωτάνε εάν συμμετέχουν Ιρανοί ή άλλοι ξένοι στις μάχες μας. Εμείς Δεχόμαστε την ε, βοήθεια της στρατιωτική της Δύσης, αλλά δεν θέλουμε στρατιωτικές βάσεις ξένες στο Ιράκ. Δεν θέλουμε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Έχουμε πολλές χώρες που είναι φιλικές προς εμάς, αλλά δεν θέλουμε να ενταχθούμε σε κάποια σφαίρα επιρροή, σε κάποιον άξονα, ούτε να αντιμαχόμεθα κάποιον άλλον και βεβαίως υπάρχει και αεροπορική κάλυψη του αγώνα μας. Όλοι οι Κούρδοι του Ιράκ είναι και αυτοί ενταγμένοι στις ε, στρατιωτικές μας δυνάμεις, είναι τμήμα των ενόπλων μας δυνάμεων και συμμετέχουν και στις δυνάμεις λαϊκής κινητοποίησης. Όλες αυτές οι δυνάμεις δρούν υπό την ηγεσία του Γενικού μας Επιτελείου. Και η συνεργασία μας δεν είναι μόνο στρατιωτική, είναι και κοινωνική, κοινοβουλευτική, διοικητική. Ο κυβερνήτης της Μοσούλης πάντα κατέχει το αξίωμά του και υπάρχει και το Επαρχιακό Συμβούλιο το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα σε ορισμένα σύνορα με την Τουρκία και με τη Συρία Ξέρετε ότι κάποιες τουρκικές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στο έδαφος της χώρας μας. Αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Το Ιράκ δεν είναι αδύναμη χώρα, βεβαίως ε, είμαστε θύμα τρομοκρατίας, αλλά και σε άλλες χώρες έχουν γίνει τρομοκρατικές επιθέσεις. Αλλά σήμερα, χάρη στις ηρωικές ένοπλες μας δυνάμεις, θα αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία. Δεν θα δεχθούμε ποτέ παρεμβάσεις τρίτων στη χώρα μας όσον αφορά την μεταβατική μας δικαιοσύνη. Τέθηκε ένα τέτοιο ερώτημα, αλλά ο συνάδελφος που το έθεσε δεν είναι πλέον παρόν. Βεβαίως υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πρέπει οπωσδήποτε η δικαιοσύνη αυτή βεβαίως να εξελιχθεί. Το θέμα αυτό το αντιμετωπίζουμε με πραγματισμό. Βεβαίως πρέπει να υπάρξουν προσωρινά μέτρα για να υπάρξουν όσο το δυνατόν ευρύτερες ε, ε, δυνατότητες προστασίας ε, του αμάχου πληθυσμού και να μην υπάρξουν παραβιάσεις του δικαίου μέσω τέτοιων προσωρινών μέτρων δικαιοσύνης. Είμαστε σε μια περίοδο φυσικά μεταβατική, αλλά και ακόμη και σε αυτή τη μεταβατική περίοδο Πρέπει να υπερισχύει το κράτος δικαίου. Πρέπει να λειτουργούν τα όργανα της δικαιοσύνης σε όλα τα επίπεδα. Και κάνουμε κάθε προσπάθεια για να το επιτύχουμε αυτό. Και στην Ευρώπη, ξέρετε, το κράτος δικαίου δεν δημιουργήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Υπήρξαν ε, φάσεις, υπήρξε μια πρόοδος προς ε, το πλήρες κράτος δικαίου και ελπίζουμε και στο Ιράκ ότι θα το επιτύχουμε αυτό, το πλήρες κράτος δικαίου ούτως ώστε να έχουμε και κοινωνική αρμονία και οικονομική πρόοδο. Τώρα, η Ρωσία και το Ιράν μας βοήθησαν. Με τους δυτικούς συμμάχους που έχουμε, προσπαθούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ε, οι χώρες αυτές μας παρέχουν μόνο αεροπορική βοήθεια. Δεν έχουν δυνάμεις επιτόπου στο έδαφος. Γιατί δεχόμεθα βοήθεια από όσους θέλουν να μας βοηθήσουν. Και οι μαχητές πέσμεργά και αυτοί συμμετέχουν. Είναι η κοινή Δεν είναι αλλοδαπή. Είναι Ιρακινοί και προασπίζουν τη χώρα τους και τις περιοχές τους. Για την προστασία των αμάχων. Πώς θα τους προστατεύσουμε από τις επιπτώσεις της επίθεσης. Το έχουμε υπόψη Έχουμε προγραμματίσει ε, μέτρα για να προστατευτούν. Με συγχωρείτε αν ήμουν ε, συνοπτικός, αλλά τέθησαν πολλές ερωτήσεις ε, και περίπλοκες. Δεν είχα χρόνο. Ήθελα να σεβαστώ το χρόνο που μου είχατε δώσει. Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, στη διάθεσή σας σε κάποια άλλη δυνατότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε και τους συναδέλφους και τους διερμηνείς και όπως βλέπετε υπάρχουν τόσες πολλές ερωτήσεις που σχετίζονται με την κατάσταση του Ιράκ. Ε, αυτό οφείλεται και στο ενδιαφέρον μας, αλλά βεβαίως και στο να λάβουμε πληροφορίες απευθείας από εσάς. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ.